δώσω τώρα ότι οι δύο ερμηνείες που αναγγέλθηκαν στην Ολομέλεια χθες για τον κανόνα 130 παράγραφος 3 και το, κανόνα, και το άρθρο 191 δεν αμφισβητήθηκαν οπότε